μέση διάταξη προβλέπει την ε, ψηφοφορία ε, με βάση την απλουστευμένη διαδικασία σχετικά με την έκθεση του συναδέλφου Ριβελίνη για την απαλλαγή του 2009. Ελεγκτικό συνέδριο. Ψηφίζουμε λοιπόν για την έκθεση με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. ψηφορία λοιπόν για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τώρα λοιπόν περνάμε. Παρακαλώ. Διαδικαστικό. Θέλω μόνο να σας πω ότι ε, δυστυχώς ε, το δικό μου το μηχάνημα δεν ε, λειτουργεί, απλά να πω ότι είμαστε παρόντες. Λοιπόν, έκθεση συναδέλφου κυρίου Ριβελίνη σχετικά με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πάλι ψηφοφορία με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. έκθεση του συναδέλφου κυρίου Ριβελίνη σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Επόμενη ε, έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή ε, και πάλι και η επόμενη είναι έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη σχετικά με το Μεταπραστικό Κέντρο των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και πάλι ψηφίζουμε για την έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφορία, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάλι για την έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη, ε, Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλίας. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή. Πάλι για την έκθεση Σταυρακάκη, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία, παρακαλώ. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή και πάλι έκθεση Σταυρακάκης ε, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Ψηφίζουμε, ονομαστική ψηφοφορία, ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται Επόμενη έκθεση Σταυρακάκης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η έκθεση. Έκθεση Σταυρακάκη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σταυρακάκης. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Σταυρακάκη. Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση Σταυρακάκης. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη, ε, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Επόμενη. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για τον Οργανισμό Εφοδιασμού της Ευρατόμ. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για την απαλλαγή πάντα του 2009 Eurojust. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για τη Frontex. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για την εποπτική αρχή του Ευρωπαϊκό GNSS, ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για την κοινή επιχείρηση άρτεμις Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη για την κοινή επιχείρηση Clean Sky. Ψηφίζουμε ονομαστική ψηφοφορία. Έκλειση ψηφοφορία. εγκρίνεται. Έκθεση ε, Σταυρακάκη ε, για την κοινή επιχείρηση, κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα. Ψηφίζουμε. Ονομαστική ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση του κυρίου ε, Σταυρακάκη, κοινή επιχείρηση Σέζαρ Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Έκθεση. Οι, οι εκθέσεις όλες αυτές του κ. Σταυρακάκη εγκρίθηκαν. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ora, del giorno... Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα της μίλησης διάταξης που προβλέπει την ε, ψηφοφορία με απλουστευμένη διαδικασία για την έκθεση ΡΑΠΚΑΙ υπεράσπιση της ε, κοινοβουλευτικής ασυλίας του κυρίου Λουίτζι Ντεματζίστρης. Ο κύριος Σιλβέστρης, είτε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω μόνο μία διευκρίνηση. Θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον η ψηφορία και η ψήφος που θα δώσουμε τώρα θα οδηγεί σε μία αυτόματη διαδικασία ή ε, είναι ένα ειδικό αίτημα του κ. Ντεματζίστρης ο οποίος ε, όλο αυτόν τον καιρό διακρίθηκε γιατί επιτέθηκε στα οικονομικά των πολιτικών και ολοκληρώνω μισό λεπτό ε, διακόπτη η πρόεδρος. Θα ήθελα να γνωρίζω αν ο ίδιος ζητάει την άρση της ασυλίας του ή αν πρόκειται για μία αυτόματη διαδικασία. Γιατί αν ο ίδιος ε, θέλει να αποφύγει την διαδικασία, η πρόεδρος διακόπτη, Κοίταξτε, εσείς ρωτάτε κατά πόσον ο κύριος Μαντζίστης ζητάει την ασυλία ή η ε, πρόκειται για μια αυτόματη διαδικασία. ποιον απευθύνεται αυτή την ερώτηση. Με ενημερώνουν ότι ο κύριος Ματζίστρης είναι εκείνος που ζητάει το αίτημα της ασυλίας. Ε, Ας προχωρήσουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε για την έκθεση. Ποιο είναι υπέρ, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι. Κατά. Η έκθεση εγκρίνεται. Έκθεση Ραπκάι, υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κυρίου Μπρούνο Γκόλνης. Ε, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, δύο λεπτά μόνο μου επιτρέπετε. Γιατί συζήτηση δεν υπάρχει, δεν μπορώ να κάνω προφορική επεξήγηση ψήφου. Με εκπλήσει πολύ αυτό κατά τα άλλα ε, με τέτοια είδους διαδικασία. Περί τίνος πρόκειται για μια πολιτική έκφραση, πολιτική έκφραση που διώκεται από τους πολιτικούς αντιπάλους Μέχρι τώρα ε, είναι διακόπτη η πρόεδρος. Θα προχωρήσουμε στην ψηφορία γιατί είχατε ήδη πολλές ευκαιρίες να εκφράσετε τη θέση σας. Όχι, όχι, δεν είχα καμία ευκαιρία να μιλήσω. Στην Ολομέλεια ποτέ. Μα και χθε, εχθέ, ε, είχα την ευκαιρία να υπερασπιστείτε τη θέση σα. Εχθέ, εν πάση αυτό δεν προβλέπεται από τον κανονισμό. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία υπέρ, παρακαλώ. Ε, να σηκώσει το χέρι. Κατά αποχές ε, η έκθεση εγκρίνεται. Έκθεση Ραπκάι άρση της ε, κοινοβουλευτικής ασυλίας του κυρίου Γκόλνης. Υπέρ παρακαλώ. Θέλετε να μιλήσετε, μα μισό λεπτό ψηφίζουμε, υπέρ παρακαλώ. Κα, αποχές κατά, εγκρίνεται. Επιθυμείτε έλεγχο, ηλεκτρονικό έλεγχο, όχι. Προχωράμε η ημερήσια διάταξη προβλέπει. Εντάξει, τότε ας ε, κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. La votazione è chiusa. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε η έκθεση. Relazione έκθεση Αρσένης ε, για την προστασία και την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής ε, του πάρκου Πρεσπών. Ψηφίζουμε υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκθεση Φράγκα Εστέβες μέτρα που λαμβάνει το κράτος ε, λιμένα για την πρόληψη της ε, παράνομης αλίας. Υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Έκθεση McCarthy για την πρόταση προσωρινών μέτρων για το πάγωμα και την γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων οφειλετών σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η εισηγήτρια έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να μιλήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σύντομα, δεν υπήρξε δυνατότητα να γίνει συζήτηση για να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου σε όλε τι πολιτικέ ομάδε που υποστήριξαν τη δική μου σύσταση και να ενημερώσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι εδώ αρχίζει η εκστρατεία του Κοινοβουλίου για να κερδίσει νέα δικαιώματα υπέρ των πολιτών που είναι θύματα απάτη. Τα προσωπικά μέτρα για το πάγωμα και τη γνωστοποίηση είναι κρίσιμα γιατί οι απαταιώνες ε, κερδίζουν, ε, δεν τιμωρούνται και τελικά ε, οι πολίτες που είναι θύματα εμπλέκονται σε μακρές δικαστικές διαδικασίες. Καταπολεμούμε έτσι λοιπόν και το οικονομικό έγκλημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Μην ξεχνάτε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ε, συνάδελφοι, τώρα πρέπει να σας διαβάσω ένα μήνυμα εκ μέρους του Πρόεδρου κ. Μπούζεκ και έχω την ευχαριστήση να σας ενημερίσω ότι σήμερα έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε τον Μπόγκταν Μπορουτσέβιτς, ο οποίος είναι Πρόεδρος της Γερασίας της Πολωνίας ε, και την Πρόεδρο ε, της ΣΕΙΜΑΣ της Λιθουανίας και την ε, κυρία Βίτβιν ε, που είναι πρόεδρος ε, της Βέτκοβα της Ουκρανίας. Οι τρεις αυτοί πρόεδροι βρίσκονται σήμερα, είναι πρόεδροι Βουλής. Κοινοβουλίου που βρίσκονται εδώ στο Στρασβούργο για μια έκτακτη συνεδρίαση Πρόεδρων Βουλής Πολωνίας, Ουκρανίας, Λιτουανίας. Και